Ένα, δύο, τρία. Καλησπέρα Σα Κυρίσω την έναρξη τη Συνόδου. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, ειδού τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ψηφοφοριών. σύσταση για τι διαπραγματεύσει ό,τι αφορά την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένου Βασιλείου. Εγκρίνεται. Διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Εγκρίνεται. Πολιτική ανταγωνισμού. Παράγραφο 1. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφο 1. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφο 2. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφο 2. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Τροπολογία 20. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Απορρίπτεται. Παράγραφος 7. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Απορρίπτεται. Παράγραφος 11. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίνεται επίσης. Παράγραφος 18. Απορρίπτεται. Παράγραφος 22. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Εγκρίνεται. Παράγραφος 27. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 28 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται επίσης. Παράγραφος 31 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 31 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 32 εγκρίνεται. Τροπολογία 5 εγκρίνεται. Η παράγραφος 34 καταπίπτει. Τροπολογία 44 εγκρίνεται. Παράγραφος 37, 36 συγγνώμη πρώτο τμήμα καταπίπτει. 36 δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Και παράγραφος 36, τρίτο τμήμα, 30, συγγνώμη, παράγραφος 37 εγκρίνεται, παράγραφος 38, τροπολογία 15 απορρίπτεται, τροπολογία 21 απορρίπτεται, παράγραφο 39 εγκρίνεται, παράγραφος 40 εγκρίνεται, 45 εγκρίνεται, παράγραφος 45, η τροπολογία 9 εγκρίνεται ομοίω. οι τροπολογίες 16 και 24 εγκρίνονται, η παράγραφο 47 καταπίπτει, μετά την παράγραφο 47, παράγραφο πρώτο τμήμα απορρίπτεται. 10, δεύτερο τμήμα απορρίπτεται, τροπολογία 11 εγκρίνεται, τροπολογία 12 απορρίπτεται, τροπολογία 17 απορρίπτεται, τροπολογία 25 απορρίπτεται, τροπολογία 18 απορρίπτεται, τροπολογία 26 απορρίπτεται επίσης. Παράγραφος 55. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 55 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Και 55 τρίτο τμήμα εγκρίνεται. 55 τέταρτο τμήμα επίσης εγκρίνεται. 57 εγκρίνεται. Τροπολογία 45 εγκρίνεται. Παράγραφος 60. Καταπίπτει. Παράγραφος 72. Εγκρίνεται. Παράγραφος 73. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 73 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 75 εγκρίνεται. Τροπολογία 13 εγκρίνεται. 82 πρώτο τμήμα καταπίπτει. 82 δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Παράγραφ, τροπολογία 30 της παραγράφου 90 απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 93 τροπολογία 29 εγκρίνεται. Τροπολογία 30 εγκρίνεται. 31 εγκρίνεται. Τροπολογία 32 εγκρίνεται. Τροπολογία 33 εγκρίνεται. Τροπολογία 34 εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 93. Πρώτο τμήμα απορρίπτεται. 22 δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. 22 τρίτο τμήμα απορρίπτεται. Τροπολογία 22 τέταρτο τμήμα επίσης απορρίπτεται. Τροπολογία 35 εγκρίνεται. Τροπολογία 36 εγκρίνεται. Τροπολογία 37 εγκρίνεται. Τροπολογία 23 απορρίπτεται. Τροπολογία 38 εγκρίνεται. Τροπολογία 27 εγκρίνεται. Τροπολογία 19 απορρίπτεται. Τροπολογία 39 εγκρίνεται. Τροπολογία 40 εγκρίνεται. Τροπολογία 41 εγκρίνεται. Τροπολογία 42 εγκρίνεται. Τροπολογία 43 επίσης εγκρίνεται. Τροπολογία 28 εγκρίνεται. Τροπολογία 7 εγκρίνεται. Στο θεωρώντα 17 ε, αυτό εγκρίνεται. Ε, τη σκέψη Β πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Ε, τη σκέψη Δ πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Ε, τη σκέψη Δ δεύτερο τμήμα επίση εγκρίνεται. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα και τώρα περνάμε στο δεύτερο γύρο τροπολογιών που ξεκινά από τις 2.30 μέχρι τις 4 παρατέταρτο. Οι ψηφοφορίες θα γίνουν με τη χρήση της ίδιας διαδικασίας. Έχετε πια εξοικειωθεί με αυτή. Τη χρησιμοποιήσαμε και το πρωί, οπότε κηρύσω την έναρξη του δεύτερου γύρου ψηφοφοριών. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι τις 4 παρατέταρτο και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν στις 6 και 4. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ένα λεπτό διακοπή και θα συνεχιστεί η Ολομέλεια.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Η ημερήσια διάταξή μας προβλέπει την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση στο χώρο Σέγγεν μετά την πανδημία της COVID-19. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους Ευρωβουλευτές ότι για τη συζήτηση αυτή δεν προβλέπεται η διαδικασία Catch the Eye, ούτε θα γίνουν αποδεκτές ερωτήσεις με τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Ο λόγος τώρα στον συντάκτη της προφορικής ερώτησης και πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, τον κύριο Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε. Αγαπητή Επίτροπε Γιώχανσον, ω πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, ε, νιώθω ιδιαίτερη τιμή που θα υποστηρίξω εδώ στην Ολομέλεια την προφορική ερώτηση για το Σέγγεν. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το Σέγγεν. Οφείλουμε να μιλήσουμε για το Σέγγεν. Έχει και γενέθλια. Στι 14 Ιουλίου του 1985, σε μια μικρή πόλη του Λουξεμβούργου, υπεγράφει μια συμφωνία και ακολούθησε το 1990 η σχετική σύμβαση και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Σέγγεν που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που βρίσκεται ισχύ. Θα πρέπει όμως να μιλήσουμε για το Σέγγεν και οφείλουμε να το κάνουμε γιατί δεν πάει και πολύ καλά η υγεία του Σέγγεν. Διακυβεύεται το ίδιο το Σέγγεν. Σέγγεν is at stake που λέμε και στα αγγλικά. Περί αυτού πρόκειται. Όσοι εργαζόμαστε στα κοινοτικά θεσμικά όργανα μερικές φορές πασχίζουμε για να εξηγήσουμε στον κόσμο τα την ορολογία την ευρωπαϊκή. Αλλά για το Σέγγεν δεν χρειάζονται εξηγήσει. Είναι το πιο πολύτιμο επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεκτημένο που μετουσιώνει τα πλεονεκτήματα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ένα εσωτερικό χώρο χωρί ε, εσωτερικά σύνορα, χωρί περιορισμού, χωρί διακρίσει μεταξύ των Ευρωπαίων. Και το χώρο αυτό τον απολαμβάνουν πάρα από 400 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες. Φαίνεται όμως ότι ο χώρος Σέγγεν ε, υπόκειται στο ενωσιακό δίκαιο, το συνοριακό κώδικα για το Σέγγεν. Πρόκειται για έναν ε, δεσμευτικό κανονισμό για τα κράτη-μέλη, που μπορεί να τον επικαλεστεί κανείς και στα δικαστήρια υπέρ της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει κάποιους όρους για την επαναφορά των εθνικών συνόρων για λόγου εθνική ασφάλεια. Βρεθήκαμε όμω σε μια πρωτοφανή κατάσταση, άνευ προηγουμένου. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία COVID-19. Εξού και το ψήφισμα που θα ακολουθήσει την προφορική ερώτηση έχει τον τίτλο το Σέγγεν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. Τι συνέβη λοιπόν με το Σέγγεν, με το χώρο Σέγγεν μετά την COVID-19. Τα κράτη-μέλη έσπευσαν να υιοθετήσουν ασυντόνιστα μονομερή μέτρα, χωρίς καν να ενημερώσουν τις υπόλοιπες χώρες, ε, επαναφέροντας τα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας τεράστιες σουρές στα σύνορα, δημιουργώντας ε, υπερβολικό φόρτο στις αστυνομικές αρχές, δημιουργώντας προβλήματα στον ανεφοδιασμό ζωτικών προϊόντων και δημιουργώντα προβλήματα και στου διασυνοριακού εργαζομένου που επίση ε, τη χάνουν προστασία από το ενωσιακό δίκαιο. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε στην προφορική ερώτηση. Και μάλιστα τα θέσαμε όλα αυτά με σαφήνεια. Πρώτον, θεωρείτε ότι τα μέτρα και οι περιορισμοί που επιβλήθησαν σέβονται τον κώδικα των συνόρων του Σέγγεν που, προτι... που κατοχυρώνει τρεις αρχές. Την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη αλλά και την απέτηση σεβασμού του δικαίου. Είναι σίγουρο ότι επανειλημμένως ε, επικαλέστηκαν τα κράτη-μέλη την εθνική ασφάλεια για το κλείσιμο των σύνορων μετά τρομοκρατικέ επιθέσει. Αλλά η δημόσια υγεία ποτέ δεν αναφέρθηκε. Για τα εξωτερικά σύνορα ναι, αλλά όχι για τα εσωτερικά σύνορα. Αυτό είναι ένα δίδαγμα που θα πρέπει να αντλήσουμε έχουμε την ανάκαμψη του Σέγγεν, γιατί έχουμε το σχέδιο ανάκαμψη. Το Σέγγεν πώ θα το ανακτήσουμε για να έχουμε απρόσκοπτη λειτουργία του και πάλι το συντομότερο δυνατόν. Και τρίτον, πώ θα μεριμνήσουμε ώστε να είναι έκτακτη έλεγχη όπως προβλέπει ο κώδικας των συνόρων και επίσης θα είναι πρόσκαιρη αυτή η έλεγχη, προσωρινή, με αυστηρό χρονικό περιορισμό. Επίσης, τέταρτον, τι πρακτικά μέτρα μπορούμε να υιοθετήσουμε για να εξασφαλίσουμε την συντονισμένη ευθύνη και την κοινή ευθύνη των κρατών μελών απέναντι σε κοινέ προκλήσεις αυτό να υπερψηφίσουμε το ψήφισμα που δίνει συνέχεια σε αυτή την προφορική ερώτηση, ευχαριστώντας φυσικά την ομάδα ελέγχου για το χώρο Σέγγεν, με πρόεδρο την Τάνια Φαγιόν. Αλλά το περιεχόμενο του ψηφίσματος είναι ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε αυτοσχεδιασμούς, δεν θέλουμε μονομερείς αποφάσεις και μονομερή μέτρα συντόνιστα. Δεν θέλουμε μια δυναμική δράση αντίδρασης του ενός κράτους απέναντι Συγγνώμη που σας διάκοψα, κύριε Αγγιλάρ, αλλά υπήρξε Το θέμα ήταν το Black Lives Matter. Φυσικά, οι ζωές των μαύρων μετράνε. Και μετράει όμως και το Σέγγεν, μας ενδιαφέρει και το Σέγγεν. Μετράει και το ενωσιακό δίκαιο. Το ενωσιακό δίκαιο μετράει ακόμη και σε περίοδο κρίσης. Ακόμη και εν μέσω της κρίσης. Και θα πρέπει το ενωσιακό δίκαιο να λειτουργεί και εν μέσω της κρίσης και να διδαχθούμε από την πείρα μας. Επίσης, το ενωσιακό δίκαιο μετράει ιδιαίτερα σε περίοδο ειρήνης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και μετά από την προφορική αυτή ερώτηση, ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα που θα ζητήσει την πλήρη επαναφορά και πλήρη ανάκαμψη του χώρου Σέγγεν. Πλήρη ανάνυψη τη υγεία του χώρου Σέγγεν, γιατί είναι το σημαντικότερο και εκτιμένο και επίτευγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Λόπε Αγγιλάρ, αγαπητέ Χωάν Φερνάντο. Και τώρα, εκ μέρου του Συμβουλίου, το λόγο έχει η Υπουργό Παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ, του τελευταίου μήνε η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε την ε, πιο σημαντική της κρίση από την ίδρυση της. Πέρα από το βαρύ τίμημα μα σε ανθρώπινε ζωέ, ε, η πανδημία του COVID-19 έχει υπονομεύσει βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού έργου, όπω η ιστορική αγορά και η ελευθερία μετακίνηση κυκλοφορίας. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο βασική προτεραιότητα ήταν να επιβραδυνθεί και να ανακοπεί η ταχεία εξάπλωση του ιού. Και έτσι πολλά κράτη-μέλη αναγκάστηκαν να πάρουν νομοθετικά και πρακτικά μέτρα τα οποία είχαν σημαντικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Και η εκ νέου εισαγωγή εσωτερικών ελέγχων θεωρήθηκε απαραίτητα από κάποια κρατημέλη τα οποία πριν από την πανδημία ήταν ε, πολύ διστακτικά για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων και σύμφωνα με τις ε, κανόνες για τους Σόγγεν η ε, εκ νέου επαναφορά των ιστορικών ελέγχων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελεί μέτρο ίστη τη προσφυγή και είναι στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Αυτό εξαρτάται και από του όρου που διευκρινίζονται του σχετικές ρήτρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακα των συνθήκων και οι, τα κάθε μέλη δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτές τις διατάξεις. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι όλοι έχουν συνεργαστεί με τις πολιτικές συνιστώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να περιοριστούν οι παράπλευρες απώλειες από την εφαρμογή των μέτρων αυτών στους πολίτες και μια σειρά ανακοινώσεων έχουν υλοποιηθεί από τα κράτη μέλη κατά προτεραιότητα για να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση και εισαγωγή ε, προϊόντων, ε, φαρμάκων, προσωπικών ειδών και σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, δυσνοριακών εργαζομένων και τον επαναπατρισμό πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη έχουν εκ παραλλήλου απαγορεύσει ε, έχουν επιβάλει περιορισμού ό,τι αφορά τι μη δικαιολογημένε ε, αφήξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη τώρα ξεκίνησαν σιγά-σιγά να χαλαρώνουν ε, τους κανόνες αυτούς σε ό,τι αφορά και την μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί μια βαθμιαία προσέγγιση και αντικατάσταση των εσωτερικών αυτών ελέγχων με άλλα μέτρα όπως ο αστυνομικός έλεγχος και έτσι τα κρατημέλη στην επικράτειά τους με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύονται να εφαρμόσουν ό,τι μέτρα χρειάζεται τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Τα πιο πολλά και οι συνδεδεμένες χώρες ε, με τον χώρο Σέγγεν έχουν άρει τους ελέγχους ε, μέχρι μάλιστα τα μέσα Ιουνίου. Οι υπόλοιπε χώρε θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του μέχρι τα τέλη του μήνα. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν, κυρίω σε ό,τι αφορά την ε, ομογενοποιημένη, αν θέλετε, άρση των μέτρων. Έχουν κινητοποιηθεί λοιπόν διάφορα ε, μέτρα χωρίς να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και όλα αυτά ε, μαρτυρούν την βασική προθυμία των κρατών να επιτρέψουν στον χώρο ΣΕ για να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την θετική ορμή με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νομικό πλαίσιο για τους ιστορικούς ελέγχους για να ξεκινήσει μια επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των συνομοθετών στο βασικό αυτό θέμα που είναι η διαφύλαξη του Σενιέν. Οποιαδήποτε λοιπόν τροποποίηση στο καθεστώς εσωτερικών συνοριακών ελέγχων θα πρέπει να ελέγχεται για να δώσει πιστικές απαντήσεις στο κοινό σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας. Θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα και ευελιξία για τα κράτη-μέλη και να μην υπάρχει περιθώριο κατάχρησης των όρων αυτών στην εφαρμογή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μπρίνιατς. Και τώρα το λόγο έχει από την Επιτροπή η Επιτροπός Γιώγανσον. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, το Σένιαν είναι ένα από τα βασικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτιμούν ιδιαίτερα οι πολίτες μας όπως πολύ σωστά τόνισε ο ε, Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ, ε, πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα έλεγα επίσης ότι όχι μόνο γιορτάσαμε την 35η επέτειο του Σέγγεν, αλλά πέρασε το Σέγγεν και μια πολύ σημαντική δοκιμή. Ε, ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντικό το Σέγγεν όσο τους τελευταίους μήνες. Όλα τα κράτη-μέλη έλαβαν ε, δραστικά μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες μας από τον ιό. Οι περισσότερες χώρες ε, Σέγγεν ε, εισήγαγαν προσωρινούς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους. Ε, μαζί με άλλα μέτρα που περιόρισαν την ελεύθερη κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα μαζί αυτά τα μέτρα βοήθησαν ώστε να σωθούν ε, δεκάδες χιλιάδες ε, ζωές, αλλά είχαν και σημαντικές, σοβαρές συνέπειες για την ελεύθερη κινητικότητα και είχαν επίσης σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Στις 15 Απριλίου φέτος, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Συμβουλίου παρουσίασαν έναν κοινό ευρωπαϊκό οδικό ε, για την άρση των μέτρων ε, για τον κορονοϊό. Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 15 Μαΐου ένα σχέδιο που παρουσιάζει μια βαθμιαία άρση μέτρων και ελέγχων των εσωτερικών συνόρων. Σε δεύτερη φάση Προσβλέπουμε και στην ε, ε, άρση των περιορισμών ε, στα ταξίδια, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης τη Δευτέρα αυτή τα περισσότερα κρατημέλη έχουν άρει τα μέτρα αυτά όπως είναι η καραντίνα μετά από κάποια μετακίνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να άρουν τους εσωτερικούς συνοριακού ελέγχους και τους περιορισμούς στην ελεύθερη κινητικότητα ε, μέσω ε, θαλάσσης ε, ξηρά και αέρος. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχουν αρθεί όλοι αυτοί οι περιορισμοί πριν ξεκινήσουμε την χαλάρωση των μέτρων που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα. Δύο έως έξι μήνες μπορούν τα κράτη-μέλη να επανισάγουν ε, ελέγχους συνοριακούς είτε σε κάποια τμήματα των συνόρων τους είτε σε όλα τα εσωτερικά τους ε, σύνορα. Ε, με διμερείς επαφές ε, με υπουργούς και με τις τακτικές ε, τηλεδιασκέψεις που έχω με τους υπουργούς και με βάση τα συμπεράσματα της ομάδας για τον κοροναϊό καταφέραμε να λύσουμε πολλά προβλήματα όπως είναι και το εύρος των, της επανεισαγωγής συνοριακών ελέγχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του κώδικα Σέγγεν. Από το 2016, έξι κράτη-μέλη έχουν επανεισάγει εσωτερικές, ε, εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους ε, κατόπιν σύσταση του Συμβουλίου ε, λόγω, για παράδειγμα, τρομοκρατικών επιθέσεων και άλλων παραγόντων. Αυτή η συνοριακή έλεγχη είχαν ε, ε, παραταθεί μέχρι ε, μέχρι και πέρσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει εναλλακτικέ λύσει ω προ του συνοριακού ελέγχου, όπω είναι η αστυνομική έλεγχη και όπω εξηγούμε στην σύσταση της 12ης ε, Μαΐου 2017 ε, μπορούν ε, να γίνονται αστυνομικοί έλεγχοι στις συνοριακές περιοχές και έτσι να αντικαταστήσουν τους συστηματικούς συνοριακούς ελέγχους. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης τροποποίηση των κανόνων διακυβέρνησης ΣΕΝΙΕΝ, ώστε η επανεισαγωγή ε, εσωτερικών συνοριακών ελέγχων να, είναι, να αποτελούν αποκλειστικά την ίστατη επιλογή. Όπως γνωρίζετε, η σχετική πρόταση έχει κολλήσει, αλλά ε, πρέπει να επανεξετάσουμε την επανεισαγωγή ε, των ελέγχων, όπως έγινε πρόσφατα, για να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Χρειάζονται πρακτικά και νομικά βήματα για να βελτιώσουμε τη ε, δυνατότητα ανταπόκρισης μας σε περιπτώσεις κρίσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πανδημιών. Θα πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ε, επέμβει μόνο σε περίπτωση ε, έμονων απειλών στα εξωτερικά σύνορα που θέτουν σε κίνδυνο την ζώνη Σέγγεν. Θέλουμε λοιπόν ε, να βρούμε απλοποιημένε και τυποποιημένε διαδικασίε που να μπορούν να εφαρμοστούν ε, υπό την πίεση των γεγονότων. Ε, θα πρέπει επίση να γίνεται διαβούλευση όσον αφορά την επανεισαγωγή και ενδεχομένω να γίνονται και συναντήσει συναντήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εμπειρίε μα του τελευταίους μήνες δείχνουν ότι αυτή η διάταξη του κώδικα Σέγγεν πολύ σπάνια χρησιμοποιείται τελικά. Το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο θα παρουσιάσω σύντομα θα είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια διαδικασία για την αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να έχουμε μια πλήρω λειτουργική ζώνη Σένιεν. Θα εξετάσουμε πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε το συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε περιπτώσει ε, επίγουσε στο μέλλον και θα ε, συλλογιστούμε και πάνω στο μέλλον του Σένιεν και θα φροντίσουμε το νομικό πλαίσιο να είναι έτοιμο για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε νέε προκλήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε στις παρεμβάσεις εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Παόλο Ραντζέλ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφυσβήτητα, το Σέγγεν είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό και εκτιμένο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Και, και παρόλα αυτά διακυβεύθηκε από την πανδημία αυτή και τέθηκε σε κίνδυνο πρωτοφανή στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη πανικοβλήθηκαν και για να προστατεύσουν τους πολίτες τους αντέδρασαν με συντόνιστο και μονομερή τρόπο, παρόλο που ήταν κατανοητό ο σκοπό τη προστασία των πολιτών. Θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και να ανακτήσουμε, να επαναφέρουμε το Σέγγεν με σεβασμό τη αρχή του συντονισμού και τη συνεργασία. Και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι εργόδει τη προσπάθειε. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συντονιστούν και να συνεργαστούν για να επαναφέρουμε το χώρο Σέγγεν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Και τώρα θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο και να το επισημάνω και στον πρόεδρο Λόπε Αγγιλάρ. Δεν είναι αλήθεια ότι ο κώδικας συνόρων Σέγγεν δεν επιτρέπει η επίκληση της δημόσιας υγείας. Γιατί μια σοβαρή απειλή της δημόσιας πολιτικής συμπεριλαμβάνει και την απειλή ε, της δημόσιας υγείας σε περίπτωση μιας πανδημίας για παράδειγμα. Η δημόσια υγεία για τα εξωτερικά σύνορα είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επιδημία ή πανδημία. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα νομότυπο λοιπόν που επικαλέστηκαν τη δημόσια υγεία τα κράτη-μέλη για αυτό που συνέβη. Σας ευχαριστώ. Σας θέλουμε παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο αγόρευση που έχετε. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Τάνια Φαγιόν. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ καταρχήν για την ε, στενή συνεργασία και τις πολυάριθμες ε, συναντήσεις που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ξέρω ότι όλοι έχουμε επίγνωση πόσο σημαντικό είναι να αναζωογονήσουμε και να ανανεώσουμε το Σέγγεν. Χωρίς ανανέωση του Σέγγεν δεν πρόκειται να ανακάμψει ούτε η ευρωπαϊκή μας οικονομία. Πρόκειται για την ε, επέτειο του Σέγγεν, την 35η επέτειο του Σέγγεν και ουδέποτε δεν είχαμε αντιμετωπίσει τόσο σοβαρή απειλή όπως σήμερα. Σε αυτή την υγειονομική κρίση διαπιστώσαμε ότι τα κράτη-μέλη έλαβαν μονομερώς κάποια μέτρα. Δεν υπήρξε κανένα συντονισμό. Έμειναν κλειστά τα σύνορα. Ο κόσμος δεν μπόρεσε να περάσει τα σύνορα, να επιστρέψει στις αιστείες του. Δεν μπορούσε να αγοράσει ιατρικό εξοπλισμό ούτε καν ε, οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας δεν μπόρεσαν να περάσουν τα σύνορα. Διαπιστώσαμε ότι ήταν τεράστια αυτή η δοκιμασία για το χώρο του Σέγγεν. Την τελευταία τετραετία είχαμε πολλέ φορέ επαναφορά των σύνορων στα εσωτερικά σύνορα χωρί νομικέ βάσει και χωρί βάσιμα νομικά επιχειρήματα. Τέτοιοι περιορισμοί και τέτοια μέτρα απειλούν το σύνολο του χώρου Σέγγεν απειλούν το σύνορο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν δικαιολογημένα αυτά τα μέτρα στη Σλοβενία, για παράδειγμα, στη Νόβα Ήταν πολύ πιο εύκολο να πάει κανείς από τη Σλοβενία στη, στο τελικό τμήμα της Σλαβαγκόριτσα από το Μάριμπορ που ήταν στην ίδια τη χώρα, τη Σλοβενία. Και όταν μιλούμε για κοινή πολιτική ασύλου θα ήθελα να πω το εξή. Αν συνδέσουμε το χώρο Σέγγεν και την επαναφορά του χώρου Σέγγεν με το θέμα του συμφώνου ε, για τη μετανάστευση και το άσυλο, θα αποτύχουμε και στα δύο θέματα. Θα πρέπει να μείνουν ξεχωριστά αυτά τα δύο θέματα. Και τα δύο ζητήματα, και ο χώρο Σέγγεν και το σύμφωνο ε, μετανάστευση και ασύλου είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να τηρηθούν και ε, την ευθύνη την έχουν τα κράτη-μέλη. Εκ μέρου του Renew Europe, το λόγο έχει ο κύριο Τουντοράκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, κυρία Υπουργέ. Διαπιστώνουμε και βλέπουμε τις δηλώσεις ε, Σούμαν και βλέπουμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα ε, και στην πράξη και τι μιλάμε για, όταν μιλάμε για αλληλεγγύη. 35 χρόνια αργότερα έγινε ένα μικρό βήμα και ξέρουμε και βλέπουμε τι σημαίνουν τα σύνορα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα 35 χρόνια. Το Σένιεν είναι μια βασική αρχή, μια βασική ελευθερία. Σήμερα όμως που αντιμετωπίζουμε την πανδημία, φάνηκαν και πάλι τα σύνορα και βλέπουμε και πάλι την Ευρώπη των ε, σύνορων και των ε, περιορισμών, χωρίς συντονισμό από πλευρά των κρατών μελών. Έκλεισαν λοιπόν και πάλι τα σύνορα και εδώ διερωτώμαστε τι ακριβώ σημαίνει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αυτή η κρίση κατέδειξε ποιε είναι οι αδυναμίε μα, αλλά και πολλά άλλα προβλήματα για του πολίτε, για τα κράτη. Και διαπιστώσαμε πόσο χρειαζόμαστε οι του δε. Θα πρέπει λοιπόν να ενδυναμώσουμε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από τα μεμονωμένα μέλη τη. και απομένει το ερώτημα του τι γίνεται με τους πολίτες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας που είναι μονίμως εκτός του Σέγγεν. Αυτό είναι η καθημερινότητά τους. Είναι όμως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ρουμανία και η Βουλγαρία αξίζουν να ζήσουν το τι σημαίνει πραγματικά η Ευρώπη για όλους. Και αυτό αποτελεί και μια έκκληση προς την Γερμανική Προεδρία για να το θέσει αυτό στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Τουντοράκη. Εκ μέρου ε, τη ομάδα ε, Ταυτότητα και Δημοκρατία, η κυρία Ταρντίνο, για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για μα είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι τα κράτη-μέλη διατηρούν την κυριαρχία για τη διαχείριση των ε, εσωτερικών του συνόρων. Ήμασταν όμω από τι πρώτε χώρε που από το ξέσπασμα της πανδημίας ζητήσαμε περιορισμούς στις μετακινήσει. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σήμερα εκπροσωπείται εδώ από την Επίτροπο Γιώχανσον, επέκρινε την επανεισαγωγή ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα και προσπάθησε να καθυστερήσει τους περιορισμούς στα εξωτερικά σύνορα κλείνοντα τα μόνο αφού η πανδημία είχε ξεφύγει του ελέγχου σε πολλέ χώρε. Αν μα είχατε ακούσει θα είχαμε μειώσει δραστικά την εξάπλωση τη πανδημία στην Ευρώπη και θα είχαμε αποφύγει την ε, εισβολή κυρίω στη Σικηλία λόγω τη εκθετική αύξηση των αφήξεων πλοιαρίων με λαθρομετανάστε. Σαν να μην μα έφταναν οι βασανιστέ που, κατέπλεψαν, που κατέπλεψαν με το πλοίο τη Καρόλα Ρακέτ. Πάντω ελπίζω τώρα να μειώσουμε δραστικά την ε, πανδημία και να να προστατεύσουμε σημαντικού ε, κλάδου τη Ευρωπαϊκή οικονομία. Όπω είναι οι μεταφορές, ο τουρισμό, οι υπηρεσίες τη φιλοξενία που υπέστησαν τεράστιες ζημιέ. και γι' αυτό δεν κουβέντα από τι άλλε ομάδε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριος που σεβαστήκατε και το χρόνο σα. Εκ μέρου τώρα των Πρασίνων, το λόγο έχει η κυρία Στρίκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Μάρτιο τα κράτη-μέλη ξαφνικά αναγκάστηκαν να λάβουν πολλά μέτρα για να καταπολεμήσουν την εξάπλωση του ιού COVID-19 και πολλά από τα μέτρα αυτά ήταν ε, σχετικά και με το κλείσιμο των συνόρων. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά δεν ε, συνάδει με ένα χώρο που υπάρχει ελευθερία κυκλοφορία και θεμελιώδη δικαιώματα και υπάρχει και η αρχή τη μη διακριτική μεταχείριση. Αποτέλεσμα λοιπόν του ότι έκλεισαν τα σύνορα είναι ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμειναν ε, εκτός της χώρας τους, δεν μπόρεσαν να πάνε στη δουλειά τους, να επισκεφθούν την οικογένειά τους, αν ήταν σε άλλη χώρα. Και βλέπουμε... Καλούμε τα κράτη-μέλη να εστιαστούν πιο πολύ σε μέτρα για την υγειονομική περίθαλψη, πιο αναλογικά μέτρα και να σιγουρευτούν ότι υπάρχει συντονισμός, κυρίως στις διασυνοριακές περιοχές, γιατί τα ιστορικά σύνορα πλέον είναι ανοιχτά. Τα εξωτερικά σύνορα είναι κλειστά όμω ακόμα. Και εδώ βλέπουμε ότι οι έντοντε άσυλο έχουν πρακτικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ε, αναζήτηση βοήθεια. Και υπάρχει και πρόβλημα επαναπατρισμού με την οικογένεια των μεταναστών. Καλούμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταπολεμήσουν αυτέ τι παραβιάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από του συντηρητικού. Η κυρία Προκατσίνη για ένα λεπτό έχει ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κρίση αυτή κατέδειξε ότι η ιδέα της Ευρώπης όπως σχεδιάστηκε πριν από πολλά χρόνια δεν ήταν επιτυχής. Το να προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, τον σχεδιασμό αυτό για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση δεν ήταν πολύ αποτελεσματικό. Ε, είχαμε, μη, είχαμε έλλειψη συντονισμού, είχαμε χάος, ενώ ε, έγινε προσπάθεια να ανοίξουν ε, τα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική κρίση. Μάλιστα, ε, είδαμε ε, να ε, αποβιβάζονται χιλιάδες μετανάστες στην Ιταλία από πλοίο που ανήκε σε μη κυβερνητική οργάνωση ενώ πέθαιναν ένα σωρό συμπατριώτες μας. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Ευχαριστώ κυρία Ντέιλι. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το κεκτημένο Σέγγεν αυτή τη στιγμή μπορεί να συνοψιστεί ω εξή. Ε, η ελεύθερη κινητικότητα είναι μια σημαντική, μια κεντρική ευρωπαϊκή αξία, εκτό ε, όταν δεν μα βολεύει, εάν είναι κανεί μαύρο, για παράδειγμα, ε, ή έχει καταγωγή που δεν μα αρέσει.